Ε, τομείς όπου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Σε περιοχέ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια για την σύνοψη αυτή. Ολοκληρώθηκε η κοινή συζήτηση και θα πραγματοποιηθεί σήμερα η ψηφοφορία. Φτάνουμε στις ψηφοφορίες. branché Καθίστε παρακαλώ Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Ρέντα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο βιομηχανικών τεχνολογικών ικανοτήτων και ερευνητικό κέντρο ε, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ε, δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού. Ε, ψηφίζουμε ε, συνολικά τις ε, τροπολογίες αρμόδιας επιτροπής υπέρ κατά αποχές, υιοθετείτε. συνεχεία, τροπολογία 11, σε εδώ δύο μέρη. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 25 υπέρ κατά άποχες υιοθετείτε. 48 υπέρ κατά άποχες διοθετείται 62 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες υιοθετείτε. δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες υιοθετείτε 159 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε 160 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 161 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχέ, υιοθετείται. 168 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 183 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ. Πάμε στην τροπολογία 186 ε, με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. Άρα, η επόμενη καταπίπτη. Όχι, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Την 184 διορθώνει η Πρόεδρος σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά της 184. Έτσι. Δεύτερο τμήμα της 184 ψηφίζουμε τώρα. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη με ονομαστική κλίση την 187D. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, στην 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Λοιπόν, 185 επαληθεύουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα. Άρχεται. Le vote Πέρας. Εγκρίνεται μεγάλη προσεφία. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 185. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο 120. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση για την 181. τη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά εποχές. Επαληθεύουμε. 182. Πέρας οφορίας. Απορρίπτεται. Ονομαστική κλίση για την πρόταση Κομισιόν. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Κυρία Ρέντα, φέρτε το λόγο. Εμπρός. Derrière. Και πίσω. Τώρα λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Σύμφωνα με τον κανόνα 59 θα ήθελα να αναπευθεί στην Επιτροπή η έκθεση αυτή για διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης Ρέντα, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Το θέμα πηγαίνει στην αρμόδια Επιτροπή για Διαθεσμικές Διαπραγματεύσεις. Περνάμε στην έκθεση ΔΕΜΟΝΤΕ, τροποποίηση του Καονισμού που αφορά την αποχώρηση του Ομένου Βασιλείου από την Ένωση. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρας προφορίας. Είναι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, η οποία ολοκληρώνεται έτσι, μετά από αυτήν την ψηφοφορία, και πάμε στην έκθεση Ντελή, τροποποίηση του Καονισμού τη Ένωση για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση την τροπολογία 25. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρα ψηφοφορία. Διοθετείτε. Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Πάμε στην έκθεση Μάισνερ λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία. Κυρία Μάισνερ, έχει το λόγο. Εμπρός. Ναι, νομίζω τώρα λειτουργεί. Συνάδελφοι, ήθελα πολύ σύντομα να σας πω ποιο είναι το θέμα εδώ. Ψηφίζουμε για την καλύτερη διάθεση των ε, αποβλήτων των πλοίων ε, στα ε, λιμάνια της Ευρώπης. Θα απαγορεύεται η απόρριψή τους στη θάλασσα, θα πληρώνεται τέλος μαζί με τα τέλη λιμανιού για να μην υπάρχει κίνητρο απόρριψης στη θάλασσα. Αυτό είναι αποφασιστική βελτίωση για τις θάλασσές μας αλλά θα μπορούν και τα σκάφη αλληλείας να παρατήθουν στα λιμάνια χωρίς επιπλέον τέλος ε, τα απορρίμματα που βρίσκουν στη θάλασσα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία και ε, προσβλέπω σε μια ευρία πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Θα το δούμε πάρα αυτά. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 117 με ονομαστική κλίση. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρας Όντω υιοθετείται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Πάμε στην έκθεση Σελίμοβιτ, παράταση τη μεταβατική χρήση μέσων άλλων τη ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασία δεδομένων προβλέπονται με τον ενωσιακό τελωνιακό κώδικα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρα φοφορία. Υιοθετείτε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό σημαίνει ότι υιοθετούμε και ολοκληρώνουμε την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Πάμε στην έκθεση Κάουφμαν, κατά πολέμηση απάτη και τη πλωστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμή πλην των μετρητών. Ψηφίσουμε τροπολογία 79 με δομαστική κλίση. Πέρα φοφορίας. Υιοθετείται η... Ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία τη αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού. Ανώτατα όρια καταλήπων για διάφορε ουσίε συμπεριλαμβανομένε και τη κλώθιανιδίνη. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. Χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία, αγαπητοί συνάδελφοι. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρα Υιοθετείτε. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Yes, now it is. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, λαμβάνω γνώση αυτού του ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου να επιβεβαιώσω ότι το σχέδιο κανονισμού ευθυγραμμίζεται με τα διαδικαστικά βήματα της απόφασης του Συμβουλίου του 1999-468 για την Επιτροπολογία καθώς και τον κανονισμό 396 του 2005. Γι' αυτό εμπίπτει στις εκτελεστικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω ότι η μόνιμη επιτροπή έχει δώσει θετική γνωμοδότηση και το Συμβούλιο ήδη έχει λάβει απόφαση να μην φέρει αντίρρηση. Λυπάμαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει το μέτρο αυτό, το οποίο βασίζεται σε ε, επιστημονική αξιολόγηση της ε, Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Έτσι, υπονομεύεται η προσέγγιση που στηρίζεται στα επιστημονικά στοιχεία. Αυτό ήθελα να πω στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε στην ψηφορία για την αντίρρηση σύμφωνα με τον αριθμό 106 του κανονισμού για γενετικό τροποποιημένο αραβό του 4114. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού για γενετικό τροποποιημένο αραβόστο μον 87 4-11. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η αντίρρηση. Επόμενη αντίρρηση πάλι σύμφωνα με το άρθρο 106. Γενικό τροποποιημένο αραβόστο BT11 ΜΥΡ 162 1507 G21. Υποχρεωμένα να τα πω κι εγώ. Με ονομαστική κλίση άρχεται. Εγκρίνεται η αντίρρηση. Και τέλο, αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού, δραστικέ ουσίε συμπεριλαμβανομένε τη θιακλοπρίδη. Με στη και πάλι άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται και αυτή. Α περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφορία έκθεση του 2008 για την Τουρκία. Έκθεση κάτι πύρη. Θα ξεκινήσουμε με την 16 με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη, δεν ήταν σαφέ, συνάδελφοι. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 5. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 2 και 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι τόσο σαφές. Ας ελέγξουμε την τροπολογία 6. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 σε τέσσερα τμήματα. Με ονομαστική κλίση το κάθε ένα. Πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3 και πάλι μονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη, δεν είμαι σίγουρη. Ας ελέγξουμε την 8. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 21 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την τροπολογία 4.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 αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά τη 10. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρωτότυπο κείμενο, Μένουμε στη κλίση, άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν επί του πρωτότυπου κειμένου. Μανομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση τη 14. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 15. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν επί του πρωτότυπου κειμένου. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Βίζα 3, πρωτότυπο κειμένο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο 6. Πρωτοποκείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Πρωτοποκείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19. Πρωτοποκείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε επί του, το σύνολο, του συνόλου του ψηφίσματος με κλίση άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Κυρία Πύρη. Vous avez demandé la parole. Έχετε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που στέλνετε σαφές μήνυμα προς το, το Συμβούλιο ζητώντας αναστολή του διαλόγου προσχώρησης με την Τουρκία επιδεικνύοντας όμως και αλληλεγγύη με του, τις δημοκρατικές δυνάμεις στην ε, Τουρκία. Αυτή είναι η τελευταία σχετική έκθεση και ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις εισηγητές ε, που πάντα καταφέρνουν να ενώνουν το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε στην επόμενη έκθεση. Βαντεκάντελάρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών ετήσια Επισκόπηση τη Ανάπτυξη για το 2019. Ψηφίσουμε επί τη 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 19 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 με κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 με κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 με κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση τώρα, τροπολογία 2. Αν θέλετε βεβαίω να ελέγξουμε για την 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, λοιπόν, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9, μονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11, μονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση τροπολογία 16 άρχεται. Le vote Πέρας. Απορρίπτεται. 17 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση για την τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με ονομαστική κλίση για το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα περάσουμε τώρα στην τελευταία έκθεση της κυρίας Χάρκιν, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, Απασχόληση και Κοινωνικέ Πτυχέ στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξη του 2019. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά προς αποφυγή λαθών άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται ψηφίζουμε λοιπόν επί του αρχικού κειμένου πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε. Για το τρίτο τμήμα λοιπόν άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μονομαστική κλίση για την 6. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Επί του αρχικού κειμένου λοιπόν, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται θεωρώ αλλά σε παληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα του αρχικού κειμένου άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε την τροπολογία 7 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Επί κειμένου παραγράφου 26, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είμαι βέβαιη, ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ είναι μικρή διαφορά, θεωρώ. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την παράγραφο 32 του αρχικού κειμένου. Πέρας. Εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση την τροπολογία 3 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση επίσης. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίσμου επιτροχικού κειμένου και πάλι με ονομαστική κλίση επί των δύο τμήματων. Πρώτο τμήμα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 41, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές Δεν είμαι σίγουρη. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα, λοιπόν. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αρχικό κείμενο, παράγραφος 45, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ετολογική σκέψη G. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για το τρίτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση τώρα. Α. Με κλίση ψηφίζουμε επί του συνόλου του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έγκρινεται. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής ψηφοφορίας. arvoisat kollegat pyytäisin teitä istuutumaan and please those who want to discuss with each other can you do it out? Όσοι θέλετε να συζητήσετε σε πηγαδάκια, να το κάνετε εκτός της αιθούσης, διότι θέλω να συνεχίσουμε τώρα την ε, συνεδρίαση. esityslistalla on ähm, De ja Guattierin mietintö. Τώρα την έχουμε την έκθεση Esther De Lange και την έκθεση Γκουαλτιέρη για τις, την ελάχιστη κάλυψη για τη, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Η κυρία Ντελάγκη, για τέσσερα λεπτά καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί ακόμα επικρατεί κάποια φασαρία στην αίθουσα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, συνάδελφοι, που καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η κυρία Ντελάνγκε έχει το λόγο. Οι υπόλοιποι καλό είναι τις συζητήσεις τους να τις κάνουν εκτός της αιθούσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που καταφέραμε να ε, σημειώσουμε μια συμφωνία σε αυτό το λεπτό πολιτικά θέμα. Είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα γιατί επηρεάζει τη σταθερότητα των χρηματαγορών και του τραπεζικού κλάδου που ακόμα είναι ευάλωτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τράπεζες έχουν ακόμα 800 δις ε, ε, ε, δανείων και πιστώσεων που δεν εξυπηρετούνται ή δύσκολα εξυπηρετούνται και αυτά επηρεάζουν πολύ επιζήμια την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και βέβαια είναι πολύ μικρότερος ο χώρος ε, για την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Και αυτό είναι εξίσου μεγάλο πρόβλημα. Είναι λεπτός ο φάκελος όμως, γιατί αυτά τα 820 δις ε, εν μέρη ε, αφορά στεγαστικά δάνεια, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε γεωργούς, ε, δάνεια τα οποία για πολλά χρόνια δίνονταν πολύ εύκολα και με ελλειπείς πληροφορίες. Και δεν έχει να κάνει μόνο αφηρημένε υποθέσεις, επιχειρήσεις και αφηρημένα ποσά. Πρόκειται για τα σπίτια του κόσμου ή τι επιχειρήσει του. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο θεωρήσαμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατεπηγόντω και με φιλοδοξία αλλά και με επιθυνότητα. Και θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει. Τι θα κάνουμε. Εκεί όπου η τράπεζα στο παρελθόν, ή μάλλον η μαλλον η εκθεση στο παρελθόν, έπρεπε να ε, μιλήσει μεμονωμένα στι τράπεζε για να αντιμετωπίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τώρα πλέον όλε οι τράπεζε είναι υποχρεωμένε ε, να ε, καλύψουν αυτόν τον κίνδυνο και ανάλογα με τον κίνδυνο της έκθεσης υπάρχει υποχρέωση 100% για τα τρία έτη ακάλυπτων δανείων, 7 έτη για τα καλυμμένα δάνεια ή 9 έτη ε, για δάνεια, για πιστώσεις που καλύπτονται ε, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Και εκεί έχουμε να κάνουμε με, τις, ε, με τα στεγαστικά δάνεια κατά βάση. Η ΕΚΤ επιπλέον έχει τη δυνατότητα, η τη δυνατότητα ανά τράπεζα να επιβάλλει επιπλέον υποχρεώσεις για την βελτίωση της κατάστασης, την επιτάχυνση της διαδικασίας. Σίγουρα αυτό θα είναι κάτι ε, βαρύ σαν πλήγμα από, για ορισμένε τράπεζε, αλλά καλύτερα να πάρουμε τώρα αυτά τα σημαντικά και σκληρά μέτρα παρά να ε, μεταθέσουμε το πρόβλημα στην επόμενη θητεία. Ε, είναι κρίμα βέβαια που αυτή η νομοθεσία θα ισχύει μόνο για, τη, για, τα, για τις νέες πιστώσεις, ενώ ε, παραμένει πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Δεν έχουμε φτάσει λοιπόν στο στόχο μας. Ο κανονισμός θα πρέπει να συμπληρωθεί και με μια οδηγία που σε αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του παρελθόντος να ε, τα απλουστεύσει ε, και κάπως να τα διευθετήσει. Και δουλέψαμε με το ίδιο, την ίδια ομάδα με τον συνεισηγητή και τους κοιόδης προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Εντό ενό έτου ε, θα περάσουμε στην υλοποίηση και στη θέση ενισχύ του κανονισμού. Το οποίο είναι δύσκολο ε, για ένα τέτοιο τόσο λεπτό φάκελο. Τα καταφέραμε και είμαστε περήφανοι. Ευχαριστώ τον συνεισηγητή κύριο Γκουαλτιέρη και του άλλου κοιόδη ε, εισηγητέ για τη συνεργασία, καθώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και την Αυστριακή και τη Ρουμανική Προεδρία. Και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα σε αυτό το δύσκολο, τεχνικό αλλά και πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, ευχαριστώ αγαπητή κυρία Ντελάγκη. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στο δεύτερο εισηγητή, τον κύριο Γκουαλτιέρη. Παρακαλώ. Τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε. Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει συζητηθεί πάρα πολύ και έχει εντοπιστεί ως ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να μειωθεί ο κίνδυνος στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο βασικός λόγος του υψηλού αποθέματος τέτοιων πιστώσεων είναι η βαθύτατη χρηματοπιστωτική ύφεση και κρίση που έπληξε πολλές ε, χώρες μετά την γενικευμένη χρηματοπιστωτική κρίση, όπου προσθέθηκαν και οι αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, λοιπόν, σε αυτή τη βασική αιτία προσθέθηκαν πιστοληπτικές ε, ε, πρακτικές χωρίς διαφάνεια, ε, χωρίς τους απαραίτητους προληπτικούς μηχανισμούς. Για αυτά τα στοιχεία έχουν υιοθετηθεί διάφορα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να επιληθεί το πρόβλημα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό παράγει μία μείωση των υψηλών αποθεμάτων αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των ΜΕΔ. Θέλω να ευχαριστήσω την Στέντε Λάγκη για τη συνεργασία γιατί χάρη σε αυτή τη συνεργασία σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώσαμε μια νομοθετική διαδικασία πολύ λεπτή. Και σταθήκαμε σε δύο βασικούς στόχους. Να ενισχύσουμε τα μέτρα με σκοπό την πρόληψη της υπερβολικής ισόρευσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και απ' την άλλη να το κάνουμε χωρίς να δώσουμε αρνητικά κίνητρα σε ό,τι αφορά τις οικονομίες γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αντίθετα τις οικονομίες, αλλά και να μην ε, πλήξουμε τους ε, Ε, γιατί θα πουλήσουν ε, τα ανοίγματα αυτά ε, και θα τα ξεπουλήσουν ουσιαστικά κάτι που είναι αρνητικό. Τι συμφωνία πετύχαμε με το Συμβούλιο. Καταρχάς, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε αυτό τον ε, μηχανισμό, τον προληπτικό μηχανισμό ασφαλείας μόνο στα νέα ανοίγματα από νέα δάνεια με βάση το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου που ζητούσε ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι λογικό, γιατί χρειάζεται μια επαρκής χρονική περίοδος για να προσαρμοστούμε στους νέους κανόνες και από λογιστική και από προληπτική σκοπιά. Δεύτερο στοιχείο. Στο κείμενο μιλάμε για την ε, συμπερίληψη στον ισολογισμό των τραπεζών και η διαφορά με την πρόταση της Κομισιόν είναι το... η διαφορά ανάμεσα στα εξασφαλισμένα ή μη ε, δάνεια μετά από δύο ή τρία χρόνια. Και θα πρέπει να δούμε τι απομείωση ε, θα φέρουμε στο, στα ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, διαγράψαμε κίνητρα πιθανώς αρνητικά και επιζήμια που υπήρχαν στην πρόταση της Κομισιόν που θα είχαν επιταχύνει την ρευστοποίηση ε, των ανοιγμάτων αυτών ανθρώπων που δεν είναι αφαιρέγγι, αλλά είναι αφαιρέγγι μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ε, και αυτό θα έχει αρνητικέ επιπτώσει και για τι μικρομέσεις επιχειρήσει, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Τελευταίο και σημαντικό όμω, θα ήθελα να αναφέρω, ένα στοιχείο το οποίο εισαγάγαμε. Υπάρχει μια προληπτική μεταχείριση πιο ευνοϊκή για εκείνα τα, ε, τα προβληματικά α, ανοίγματα που έχουν α, αγοραστεί σε δευτερογενείς αγορές και να προστατεύσουμε πιο πολύ τον καταναλωτή και όλους τους άλλους οφειλέτες, αυτή στιγμή αυτή η, αυτά τα ιδρύματα υπόκεινται σε σοβαρούς ελέγχους και ρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο κείμενο, θα μπορούσα να πω συμπερασματικά, και μας επιτρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα εμπρός, ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος του τραπεζικού τομέα και να αποφύγουμε παράλληλα αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στους καταναλωτές και γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους σας να στηρίξετε το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκουαλτιέρη. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Ντομπρόφσκης. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ντελάνια, κύριε Γκουαλτιέρη, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ που αναλάβατε τις εργασίες πάνω στο θέμα αυτό πέρσι με ισχυρή αίσθηση ε, αφοσίωσης και έχουμε εργαστεί τα τελευταία χρόνια εντατικά για να μειώσουμε τον κίνδυνο και να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τομέα τραπεζών. Με την ε, συγκεκριμένη πρόταση ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα των μη εξυπηρετώμενων δανείων, ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Μετά από την ε, οικονομική κρίση είδαμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Είδαμε ότι όταν υπάρχει αυξημένος ε, βαθμός κινδύνου και ε, εάν δεν αντιμετωπιστεί εν καιρός, αυτό επιφέρει κίνδυνο για το σύνολο της οικονομίας. Συνεχίζει να είναι υψηλό το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ε, δεν μπορεί να ε, θεωρούμε δεδομένη την ε, αύξηση του ΑΕΠ που έχει οδηγήσει στην πρόσφατη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τους κινδύνους για να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε να αποφύγουμε την υπερβολική συσσόρευση ε, των ε, μη εξυπηρετούμενων ε, ανοιγμάτων χωρίς επαρκή κάλυψη των απολειών. Και γι' αυτό καθορίζουμε ένα μέγιστο επίπεδο και η πρόταση αυτή αποτελεί προσθήκη στα υπάρχοντα εργαλεία εποπτείας. Ο προληπτικός μηχανισμός ασφαλείας ε, αποτελεί σημαντικό τμήμα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Αλλά η εργασία μας πάνω στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν ε, είναι ακόμα ολοκληρωμένη. Ο προληπτικός μηχανισμός ασφαλείας είναι τμήμα μιας δέσμης μέτρων και χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα και γι' αυτό σας καλώ σύντομα να εγκρίνετε την πρόταση αυτή για να προχωρήσουμε στις δευτερογενείς αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περνάμε στις πολιτικές ομάδες. Πρώτα από το ΕΛΚ, ο κύριος Γκέρολτ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, κάνουμε ουσιαστικά μια συζήτηση για την ε, πολιτική λιτότητα και τη σχέση μεταξύ των μελών. Δεν είμαι ο μοναδικό που έχει την εντύπωση ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και οι συνέπειέ τη έχουν πλήξει σοβαρά την ενότητα στην ε, Ευρώπη και ότι αυτά τα πλήγματα δεν έχουν ακόμα ε, επουλωθεί πλήρως. Ο τροπικός ταμέα ε, ζημιώθηκε πολύ σε αυτό το πλαίσιο και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και στου Ευρωπαίου πολίτε. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πολύ σημαντικά για την γενικότερη ευημερία γιατί τελικά και αυτός είναι και ο σκοπός ε, της ε, χρηστής ε, λειτουργίας του χρηματοπιστικού συστήματος. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν να επωφεληθούν των θετικών εξελίξεων στην οικονομία. Δεν είναι μόνο οι τράπεζες βέβαια, αλλά και τα άτομα που πρέπει να αποφεληθούν. Γι' αυτό, εξετάζοντας την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως αναπόσπαστο τμήμα ε, αυτής της διαδικασίας. Μπορούμε λοιπόν ε, να εξετάσουμε με ρεαλισμό το θέμα αυτό στο μέλλον. Σε χαίρον λοιπόν τους εισηγητές επειδή βρήκαν μια ισορροπημένη προσέγγιση σε πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ωστόσο βλέπουμε ότι προκειμένου να διασφαλίσουμε την ε, επιτυχία αυτής της πρότασης πρέπει παρόλα αυτά ε, να αποδεχθούμε και το πικρό χάπι της χρηστής ε, ε, διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Δεν θέλουμε ε, στασιμότητα, θέλουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές ε, λιτότητας ε, δεν αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένων κακών πολιτικών, αλλά ανεύθυνων πολιτικών που υλοποιήθηκαν από αδύναμες και αφιλόδοξες κυβερνήσεις για πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γκέρχολτ. Νίνα Γκίλ από... Νίνα Γκίλ τους Σοσιαλιστές για δύο λεπτά. Να συγχαρώ τους οι συγητέ, ε, τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη και την Έστερ Ντελάνγκ. Τα ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν κληρονομιά από την τελευταία οικονομική κρίση και μία δεκαετία μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μειώσει αποτελεσματικά τα επίπεδα. Γι' αυτό απαιτείται δράση για να αποτρέψουμε μία παρόμοια κατάσταση στο μέλλον. Από το 2015 και μετά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν ε, μειωθεί από το 1 τρισεκατομμύριο μόνο κατά 400 δισεκατομμύρια και αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη ζώνη του ευρώ. Ε, πρέπει λοιπόν οι τράπεζες ε, να καθαρίσουν ε, τους ισολογισμούς τους και γι' αυτό επικροτώ το βελτιωμένο κείμενο προϊόν του τριμερούς διαλόγου, διότι περιέχει διατάξεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και σημαίνει ότι θα μειώσουμε τις δυνάμει αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ενώ έχει μειωθεί ο κίνδυνο στον τομέα των τραπεζών σημαντικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσεγγίζει κάπως περισσότερο την Τραπεζική Ένωση, τρεις σημαντικέ μετερρυθμίσεις απαιτούνται ακόμη για να γίνει πιο ανθεκτικός ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε ένα αποφασιστικό βήμα προ ένα ε, πανευρωπαϊκό ε, καθεστώ για τι καταθέσει για να προστατεύσουμε του καταθέτε. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Είναι κρίμα που η δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου μπλοκάρει το θέμα αυτό για ιδεολογικού λόγου και ελπίζω το επόμενο Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα. Δεύτερον, η βιώσιμη χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι κανόνα και όχι η εξαίρεση. Και καθότι οι τράπεζε συνεχίζουν να είναι η βασική χρηματοδοτική πηγή τη ευρωπαϊκή οικονομία, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα πρόσφατα βήματα που έχουμε αναλάβει στην δέσμη για την βιώσιμη οικονομία ε, με κάνει να θέσω την ερώτηση στην Κομισιόν. Πώς θα φροντίσετε οι τράπεζες να αναλάβουν την ευθύνη αυτή. Και δεδομένων των ε, τεράστιων επιπτώσεων ε, στην οικονομία και στους φορολογούμενους ε, της τελευταίας κρίσης, δεν μπορούμε να έχουμε